Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμότατα μετά από το διάλειμμα που είχαμε μεταξύ της Συνόδου Ολομέλειας του Στρασβούργου και της σημερινής συνεδρίασης και θα περάσω στο καλωσόρισμα των καλεσμένων μας. Αλλά πρώτα κάποια τυπικά ζητήματα. Καταρχήν να μεταδίδεται από το διαδίκτυο απευθείας η συνεδρίασή μας και όπως ξέρετε στις 5 ε, ώρα το απόγευμα θα αλλάξουμε αίθουσα γιατί θα μεταβούμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γυναικών και ε, Ισότητας των Φίλων. Εκεί θα μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Ευτυχώς η δεύτερη αυτή αίθουσα στην οποία θα μεταβούμε είναι πολύ κοντά, είναι στον πρώτο όροφο, στο ίδιο ακριβώ ύψο. Θα κατεβούμε απλώ δύο ορόφου. Ελπίζω να μην έχετε πρόβλημα με την ημερήσια διάταξη, την εγκρίνουμε και περνάμε στο κύριο θέμα της απόψινής μας συνεδρίασης που είναι η δημόσια ακρόαση με θέμα το ρόλο της γεωργίας συντήρησης στην αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Το θέμα αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά μια νέα προσέγγιση ζωτική σημασίας για το οικοσύστημα. Από βιολογικής απόψης δηλαδή, η νέα αυτή προσέγγιση είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε η γεωργία μας να είναι πιο αποδοτική και ταυτόχρονα πιο φιλική προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα πιο φιλική προς τα εδάφη. Επίσης θέλουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους φυσικούς πόρους, καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής και περισσότερα αποτελέσματα και καλύτερη απόδοση. Οι καλεσμένοι μας είναι εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί, από πολύ γνωστά πανεπιστήμια. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την κυρία Πάολα Τριβίνιο Ταράδας, που είναι ε, project manager ε, Ομοσπονδία, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργίας Συντήρηση και επίσης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβας. Καλώ ήρθατε κυρία Τριβίνια Ταράδας. Δεύτερη εμπειρογνώμων είναι η κυρία Τζούλια Κούπερ από τη Σχολή Γεωργίας Τροφίμων και Ανάπτυξη Πέθρου από το Πανεπιστήμιο του Νιου Κάσλ. Είναι επικεφαλής ερευνήτρια στην επιστήμη του εδάφους και στην οργανική ελάχιστη άρρωση. Άλλη εμπειρογνώμη είναι μια ερευνήτρια πανεπιστημιακή, πανεπιστημιακή, κυρία Τορεμότσα, από το Πανεπιστήμιο Παύλο Δολαβίντε της Εβίλη, που ασχολείται με την έρευνα σε αγροοικολογικά θέματα, βιολογική γεωργία και τις κλιματικές αλλαγές. Και τελευταίος ε, εμπειρογνώμονα μα είναι ο κύριος Μολίνα Φάμπρα, Καθηγητή γαστρονομίας ε, στο Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάθε καλεσμένος εμπειρογνώμονας δικαιούται δεκάλεπτο χρόνο και μετά τις δύο πρώτες παρουσιάσεις θα προβλέψουμε λίγο χρόνο για υποβολή ερωτήσεων και κάποια συζήτηση με τις απαντήσεις από τους εμπειρογνώμονες. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις σας. Ε, γι' αυτό και σας καλέσαμε σήμερα. Οπότε θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Τριβίνο. Θέλουμε παρακαλώντας να μας συγχωρέσει για την ε, μικρή αυτή καθυστέρηση στην άρεξη της συνεδρίας αλλά Δευτέρα είναι αναμενόμενο ήταν κάτι τέτοιο. Κυρία Τριβίνια Ταράδας, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργία Συντήρηση νιώθει ιδιαίτερη τιμή που μέσω μου εκπροσωπείται σε, στη σημερινή ακρόαση με θέμα τη διαφύλαξη της υγεία του εδάφους ως βασικό στοιχείο, κεντρικό σημείο της ε, γεωργικής και περιβαλλοντικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, αλλά στο κανάλι 3 ακούμε τη ρουμανική διερμηνία, λέει ο κύριος Ταραμπέλα. Πρεσεντίντα, άκουσα. Ε, δεν είναι και πολύ μακριά τα γαλλικά από τα ρουμανικά. Δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα για να μην καταλαβαίνετε ρουμανικά, κύριε Ταραμπέλα. Είναι οικίες αυτές οι γλώσσες. Μουτσουμέσκ, λέει. Εντάξει, διορθώθηκε το πρόβλημα, Μα έκανε νεύμα ο κύριο Ταραμπέλα. Έχετε το λόγο, κυρία Ταράδα. Λαμπρά. Ο κύριο Άγνιο. Ναι, και μιλάμε για τη διερμηνία. Εγώ έχω βάλει στο, στο 9, στο full τον ήχο και φοράω και το ακουστικό μου, αλλά παρόλα αυτά δεν ακούω. Μήπως θα μπορούσε λοιπόν ο Άγγλος Δερμηνέας να μιλάει λίγο πιο δυνατά για τον ακούω, γιατί το έχω βάλει στο τέρμα. Και παρόλα αυτά δεν ακούω. Εντάξει, μετά αυτές τις παρατηρήσεις νομίζω ότι είμαστε εντάξει με τα τεχνικά και να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Τριβίνιο. Καλησπέρα σας και πάλι. Όπως είπα, είναι μεγάλη τιμή για την Ομοσπονδία μας, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργία Συντήρησης, να εκπροσωπείτε εδώ και να μιλά υπέρ ε, του γεωργικού εδάφους ε, που βρίσκεται στο επίκεντρο της γεωργικής πολιτικής αλλά και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργίας Συντήρησης ιδρύθηκε στο 1999 εδώ στις Βρυξέλλες, απαρτίζεται από 14 εθνικές ενώσεις ε, και μάλιστα προσπαθούμε σε όλες αυτές τις εθνικές ενώσεις να προωθήσουμε την βιώσιμη χρήση του εδάφους από τους γεωργούς. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε λίγο ε, το βαρύτατο τίμημα που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Κοινωνία για την υποβάθμιση του εδάφους. Στα αριστερά βλέπουμε τις απειλές που υφίσταται το έδαφος ε, από την θεματική στρατηγική για το έδαφος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα η δική μας Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συνέβαλε από το ε, μέχρι το 2006 στο έργο αυτό και βλέπουμε ε, κάθε φαινόμενο τι ετήσιο κόστος έχει για την υποβάθμιση του εδάφους. Και αν προσθέσουμε όλα αυτά τα ποσά, φτάνουμε στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το κόστος που καταβάλουμε, το τίμημα που καταβάλει η κοινωνία μας για την υποβάθμιση του εδάφους. Και μάλιστα πέρυσι ε, στις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις των άμεσων ε, αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις ε, της ΚΑΠ αυτό το ποσό περίπου καταβάλαμε. Βλέπετε τις φωτογραφίες και θα ήθελα να, να παρακαλώ να μην έχει αυτό το χρώμα το νερό που βλέπουν τα παιδιά μας να κυλάει στα ποτάμια μας. Γιατί αυτό το χρώμα οφείλεται στη διάβρωση, στην υποβάθμιση του, του εδάφους και στην υποβάθμιση των τροφίμων που καλλιεργούνται στο έδαφος αυτό. Πού οφείλεται λοιπόν αυτή η διάβρωση του εδάφους, κυρίως στην εντατική ε, άρρωση, γιατί αυτά τα εντατικά οργώματα υποβαθμίζουν το έδαφος, το διαβρώνουν, καταστρέφουν τη δομή του και αφήνουν ένα πολύ ευάλωτο έδαφος, ένα έδαφος που είναι επιρρεπέ στη διάβρωση. Και εδώ έχουμε πολύ εντυπωσιακέ ε, συγκλονιστικέ ε, φωτογραφίες διάβρου εδάφους, μάλιστα όχι μόνο από την Ευρώπη, σε μονοετή καλλιέργειε, αλλά και σε, πολυ... σε βλέπουμε πως ε, έχουν μείνει γυμνές οι ρίζες δέντρων και επίσης έχουμε αριστερά μία ε, άρχουσα τέτοια διάβρωση που όμως επίσης είναι απειλητική και μπορεί να μας οδηγήσει μετά από λίγα χρόνια στις φωτογραφίες της δεξιάς πλευράς. Επίσης θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι τη σήμερα ημέρα η Γεωργία με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι η ε, υπεύθυνη για το 10% περίπου των αερίων του θερμοκηπίου. Γνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι όλες αυτές οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου θα μπορούσαν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό χάρη στη χρήση καλών γεωργικών πρακτικών και χάρη στην εφαρμογή αυτών των πρακτικών της γεωργίας συντήρησης. Με τον περιορισμό ή τη μηδενική άρρωση έχουμε ε, μεγάλο περιορισμό του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, ε, αν αποφύγουμε το όργωμα, θα περιορίσουμε και την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων. Επίσης έχουμε μία στασιμότητα, μία αποτελμάτωση των ε, εσοδιών, των συγκομιδών τα τελευταία χρόνια. Κάτι που θα δημιουργήσει ακόμη, προκλή, ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις στην παραγωγή, όπως μας λέει η ΚΙΦΑΟ. Οπότε έχουμε καθήκον και υποχρέωση να βρούμε μια πολύ πιο βιώσιμη προσέγγιση για τη γεωργία μας. Γιατί δεν θα πρέπει μόνο να αυξήσουμε τη γονιμότητα του εδάφους, αλλά να τοποκριθούμε και στις προκλήσεις της παραγωγής και να αυξήσουμε τη γεωργική παραγωγή για να καλύψουμε τις ανάγκες. Εδώ θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τις βασικές, τις θεμελιώδεις ε, και αλληλένδετες αρχές της γεωργίας συντήρησης. Γιατί δεν αρκεί ε, μεμονωμένα να εφαρμόσουμε μία από τις τρεις αρχές, θα πρέπει σωρευτικά να εφαρμόσουμε και τις τρεις αυτές αρχές στα χωράφια για τη γεωργία συντήρησης. Λοιπόν, άμεση σπορά καταρχήν, χωρίς προηγούμενη άρρωση. Έτσι θα παραμείνει το περιεχόμενο στο έδαφος, δεν θα απεμπλουτιστεί και μάλιστα θα αυξηθεί η παρουσία οργανικής ύλης στο έδαφος. Επίσης θέλουμε κάλυψη του εδάφους, γιατί με την κάλυψη του εδάφους θα περιοριστεί αυτή η ροπή προς την υδρολογική και την αιωλική διάβρωση και επίσης ε, θέλουμε άμυψη σπορά, διαφοροποίηση ε, και στις μονοετής αλλά και στις πολιετές καλλιέργειες. Είναι σημαντική η αμύψη σπορά, γιατί έτσι μόνο θα ενισχύσουμε τις θετικές συνέργειες μεταξύ των διαφόρων καλλιεργειών. Ένα για παράδειγμα, έχουμε ένα ψυχανθές, που θα δεσμεύσει το ατμοσφαιρικό άζωτο, θα το κρατήσει στις ρίζες, ώστε στην επόμενη καλλιέργεια θα περιοριστεί η, ανάγκη για ε, αζωτούχα λιπάσματα. Αυτέ είναι οι τρει βασικέ αρχέ τη γεωργία συντήρησης που θα αυξήσουν αμφισβήτα και την ποιότητα του ύδατος και την ποιότητα του εδάφου, θα αυξήσουν τη γονιμότητα του εδάφους θα ενισχύσουν τη δέσμευση του άνθρακα στο έδαφος πολύ σημαντικό σημείο για τις κλιματικέ αλλαγέ, και επίσης λειτουργεί το σύστημα αυτό σε όλα τα αγροσυστήματα. Δηλαδή και για τα μονίμως ε, πάγια εδάφη του Καναδά, αλλά και σε ε, εδάφη που λαμβάνουν ε, πλούσιες βροχοπτώσεις κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι ένα σύστημα που προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε εδάφους. Αυτές λοιπόν οι βασικές αρχές της γεωργίας συντήρησης ε, είναι απόλυτα συμβατές και με άλλα μέτρα χρηστών γεωργικών πρακτικών που ήδη έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για παράδειγμα, ολοκληρωμένη στρατηγική κατά των επιβλαβών οργανισμών και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια πολύ πιο βιώσιμη και αηφόρο γεωργία που θα στηρίζεται στην ε, ε, στην μέγιστη αξιοποίηση των γεωργικών ισρών και σε μια πιο ασφαλή χρήση των ισρών αυτών. Για να διευκρινίσουμε λοιπόν ε, τις διαφορές γεωργίας συντήρησης και συμβατικής γεωργίας. Με τη συμβατική γεωργία ουσιαστικά τροποποιούμε το περιβάλλον. Με το όργωμα δηλαδή, με την άρρωση, αλλάζουμε το περιβάλλον για να το ετοιμάσουμε για τη σπορά. Ενώ στη γεωργία συντήρησης, χάρη στα νέα φυτά και τεχνολογία, προσαρμοζόμαστε στο μέσο που έχουμε, δηλαδή στο συγκεκριμένο έδαφο, χωρί να το επηρεάζουμε να το διαταράσουμε με την άρρωση. Κοιτάξτε μερικέ φωτογραφίε ε, από την Ευρώπη, Γεωργία συντήρηση, είτε με καλυμμένε καλλιέργειε, προστατευτικέ δηλαδή, ή με τις υπόλοιπε καλλιέργειε που βλέπετε στην οθόνη. Οπότε, αν καταφέρουμε πριν τη σπορά να έχουμε κατά λιγότερο του 30% καλυμμένο εδάφου, ε, ε, παρεμποδίζουμε κατά 90% τη διάβρωση και κατά 30% την απορροή του νερού. Την απώλεια νερού δηλαδή από το έδαφο. Και μάλιστα η γεωργία συντήρηση λειτουργεί σε πολλέ χώρε με διαφορετικέ καλλιέργειε, σε διαφορετικά συστήματα, όχι μόνο στα, στις καλλιέργειες του χειμώνα, αλλά και στι αερινέ καλλιέργειες. Έχουμε εδώ την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, εδώ τη Ισπανία, ε, με ελαιούχους σπόρους, με βιομηχανικέ επίση καλλιέργειε. Και αυτό που σα είπα προηγουμένω για τι. Ε, ε, μόνιμες καλλιέργειες, έχουμε επίση καλυμμένα εδάφη. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μία κάλυψη ε, με χλώη, γιατί μια τέτοια προστατευτική καλλιέργεια και ε, φρενάρει τη διάβρωση, αλλά και περιορίζει την απώλεια ύδατος από το έδαφος. Και μάλιστα, επειδή ακριβώ με την γεωργία συντήρηση δεν διαταράσουμε την ισορροπία του εδάφου, επιτρέπουμε στου μικροοργανισμού του εδάφου να παραμείνουν ε, στο έδαφος και μάλιστα να αυξηθούν. Έτσι ενισχύουμε τη βιοπικιλότητα του εδάφους. Κάτι που θα ε, επηρεάσει θετικά όλη την διατροφική αλυσίδα. Όχι μόνο το έδαφος, αλλά και τα τρόφιμα που θα παραχθούν σε αυτό το έδαφος, γιατί βελτιώνεται η επικονίαση και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε ένα απλό παράδειγμα του ίδιου χωραφιού με την ίδια πλαγιά, με καλλιέργεια αραβοσίτου, την ίδια καλλιέργεια δηλαδή, στα αριστερά βλέπουμε ε, μετά από έντονες βροχοπτώσεις ότι όχι μόνο χάσαμε μερικά φυτά, αλλά χάσαμε και το έδαφος που έχει πάθει καθίζηση. Και σίγουρα ε, αυτό επηρεάζει τον Γεωργό και δεν τον ικανοποιεί καθόλου, γιατί χάνει και γονιμότητα το έδαφος, αλλά χάνει και ποιότητα το έδαφος με τέτοιες πρακτικές. Και εδώ βλέπετε μερικά παραδείγματα από ένα πρόγραμμα που κέρδισε ε, το πρόγραμμα του καλύτερου περιβαλλοντικού προγράμματος στην Ανταλουσία, το Life ε, Sin Agri Carbon. Αυτό είναι το σχέδιο. Και μάλιστα συνεχίζουμε από κοινού με άλλα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, Life ε, για το κλίμα, που επίσης τρέχουν σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως βλέπουμε και κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ της ε, γεωργίας συντήρησης και της συμβατικής γεωργίας βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο έχουμε 56% αύξηση της δέσμευσης ε, άνθρακα χάρη στη γεωργία συντήρηση σε σχέση με τη συμβατική γεωργία. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, κατανάλωση ενέργειας. Έχουμε όχι μόνο μείωση τη κατανάλωση ενέργεια, αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Είχαμε λοιπόν μείωση κατά 19% τη χρήση ενέργειας στις τρεις ε, καλλιέργειε που εφαρμόστηκε αυτό το σχέδιο, αυτό το project. Και αυτό θα έχει σημαντικά ωφέλη και για τον ε, γεωργό, γιατί μειώνεται το κόστος παραγωγής στις καλλιέργειες αυτές και στις τρεις αυτές καλλιέργειες που είδαμε, «Σύτο», ηλιοτρόπιο και ψυχανθή, είχαμε μείωση του κόστου στη γεωργία συντήρηση σε σχέση με τη συμβατική γεωργία. Επίση θα ήθελα να σα δω από πού προέρχονται όλα αυτά, πότε ξεκίνησα, γιατί είναι σχετικά πρόσφατα, στη δεκαετία του 30 στην Αμερική, με τι ανεμοθύελες που είχαμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, αναζητήθηκε ένα τρόπο και κάποιε τεχνικέ πρακτικέ για να μπει ένα τέρμα στην νεολική διάβρωση του εδάφου. Σήμερα έχουμε φτάσει στα 160 εκατομμύρια εκτάρια στον κόσμο στον κόσμο, στην Ευρώπη δεν έχουμε ούτε 4 εκατομμύρια εκτάρια, ε, που είναι και πόδις καλλιέργειες και ε, πολιετής καλλιέργειες, ετής και πολιετής. Επίσης, ε, διαπιστώσαμε ότι η Γεωργία Σιδηρής ανταποκρίνεται κάλλιστα στις τωρινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και σε ό,τι αφορά τη γονιμότητα του εδάφους, βελτιώνεται η γονιμότητα του εδάφους με τη γεωργία συντήρηση, αλλά συμβάλλει και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και μάλιστα αναγνωρίστηκε από τη ΦΑΟ ως έξυπνη γεωργική πρακτική για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αναγνωρίστηκε και για, τους, για μερικούς από τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης και επίσης ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη γαλλική πρωτοβουλία 4 επί 1000, την πρωτοβουλία 4 επί 1000 του κόπου 21 γιατί ακόμη και μικρή δέσμευση ε, άνθρακα, τέσσερα της μπορεί να ε, βελτιώσει κατά πολύ τη γονιμότητα του εδάφους και επίσης να μειώσει την θέρμανση του πλανήτη, ώστε να μην υπερβούμε τη θέρμανση ε, πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου, που είναι και ο στόχος. Επαναλαμβάνω, η γεωργία συντήρησης έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει τη βάση της μελλοντικής γεωργικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για τις άμεσες πληρωμές, αλλά και για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για το δεύτερο πυλώνα, για τις άμεσες πληρωμές, γιατί βλέπουμε ότι με το greening, αυτό το πρασίνισμα της γεωργίας, στηρίζουμε τέτοιες γεωργικές πρακτικές που θα μετριάζουν τις κλιματικές αλλαγές και φυσικά στα πλαίσια της ανάπτυξης υπαίθρου χρησιμοποιούμε τη γεωργία συντήρησης για να καλύψουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Γεωργός κατά την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Θα ήθελα επίσης δημοσίως εδώ να ευχαριστήσω τις 140 υπογραφές που συγκεντρώσαμε για το καλοκαίρι για τη διακήρυξη υπέρ της Γεωργίας Συντήρησης. Επιτέλους αναγνωρίστηκε αυτό το σύστημα της Γεωργίας Συντήρησης, ο σύστημα που βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους, περιορίζει τη διάβρωση και μετριάζει, συμβάλλει στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Και σε αυτή τη τελευταία διαφάνεια διαβάζεται ποια είναι τα ωφέλη τα γεωργικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά από την γεωργία συντήρησης. Και μάλιστα τα έχω βάλει σε μία μνήμη USB που περιέχει βάση δεδομένων με επιχειρήματα, επιστημονικά επιχειρήματα που αποδεικνύουν και με επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις, όλα αυτά τα ωφέλη της γεωργίας συντήρησης. Και μάλιστα εκτός από τα επιστημονικά άρθρα έχετε και κάποια επιστημονικά και τεχνικά δελτία και κάποια βίντεο. Αυτά τεκμηριώνουν όλα αυτά που είπα για τα ωφέλη της γεωργίας συντήρησης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην δεύτερη πυρογνώμονά μας από το Πανεπιστήμιο του Νιου Κάσιλ, την κυρία Τζούλια Κούπερ. Και σας θέλω παρακαλώ να μην ξεπεράσετε και εσείς το δεκάλεπτο. Okay. Thank you very much for inviting... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με καλέσατε να σας μιλήσω και εγώ για αυτή την ακρόαση σχετικά με την γεωργία συντήρησης. Και θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η πόλο. Και θέλω να σας πω ότι σαφώς και είμαι επιφύλακτα υπέρ της γεωργίας συντήρησης. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποιες προκλήσεις και υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να τους έχουμε κατά νου ε, εξετάζοντα τον ενδεχόμενο να προάγουμε την ε, γεωργία στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πάλα είπε, μίλησε ήδη για τη γεωργία αυτή. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για την ε, διαταραχή του εδάφους. Ε, ε, δεν πρέπει αυτό να το εξετάσουμε περαιτέρω. Τουλάχιστον στο κάλυμα του εδάφους θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε και τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους. Να έχουμε κατά νου το βιολογικό όργωμα και να έχουμε επίσης κατά νου ότι Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να γίνει το όργωμα χωρίς να πρέπει να παρέμβουμε απαραίτητα μηχανικά. Γιατί όταν παρεμβαίνουμε μηχανικά διαταράσσουμε κατά κάποιον τρόπο το έδαφος. Και εδώ έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θα θυμάστε ότι είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο έναν πρωτοπόρο γεωργό ο οποίος ε, ε χρησιμοποίησε τη γεωργία συντήρησης. Ε, ίσως να μην βλέπετε ακριβώς το τι θέλουν να σας δείξω. Ε, αυτά, αυτή η εικόνα είναι πίσω από τη δική του τη γεωργική εκμετάλλευση. Βλέπετε την επιφάνεια του εδάφους, ε, προστατεύεται το έδαφος ε, από την απορροή, όπως είπε και η, η Άρα δηλαδή φυλάσσουμε τα οικοσυστήματα, ε, βελτιώνουμε την διείσδυση του εδάφους και τη συγκράτηση του εδάφους ε, και προσπαθούμε να αποφύγουμε την διάβρωση. Όλα αυτά αποφέρουν ωφέλη. Ε, ο τρίτος πυλώνας είναι η διαφοροποίηση της σποράς. Δεν χρειάζεται να επιμείνω σε αυτό. Το γνωρίζετε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ποικιλία. Άρα δηλαδή βασιζόμαστε στην ποικιλομορφία των καλλιεργιών. Βασιζόμαστε λοιπόν σε, πιο, σε μεγαλύτερη βιοπικιλότητα, ε, γι' αυτό οφείλουμε να σπάμε τους ε, κύκλους ε, των παρασίτων και των ζυζανίων. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες που μπορούν να βοηθήσουν ε, για να διαφυλαχθεί το έδαφος. Αυτά που βλέπετε είναι βασικοί οι πυλώνες και τώρα θα ήθελα να περάσω σε κάποιες θεωρίες και σε κάποιες αρχές γιατί όλα αυτά πρέπει και μπορούν να λειτουργήσουν. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις καταρχήν όσον αφορά την αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών. μελετών. κατά πολύ οι ε, ορισμοί, ε, το μειωμένο, το ελάχιστο όργωμα, το μηδενικό όργωμα. Αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με την γεωργία συντήρηση. Πρέπει λοιπόν όταν εξετάζει κανεί μελέτε, να έχει κατά νου να προσπαθεί να δει τι είδου όργωμα χρησιμοποιείται. Και οι άνθρωποι που τάσσονται υπέρ τη ε, ε, γεωργία συντήρηση επιθυμούν κυρίως το μηδενικό όργωμα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς μελέτες ε, οι οποίοι κάνουν πρακτικές δοκιμές. Πολλές φορές οι μελέτε μελέτες εξετάζουν μόνο το όργαμα και όχι την άμυψη σπορά ή τη βιοπικιλότητα. Είναι λοιπόν δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα για τους διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται ε, για να δούμε ε, πώς μπορούμε να περιορίσουμε το όργαμα από την αναστροφή, τη βαθιά αναστροφή. Ε, η βαθιά αναστροφή είναι αυτό το οποίο θεωρούμε ως το παραδοσιακό όργωμα. Μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς τις επιστημονικές μελέτες για να καταλήξει ε, στο ποια είναι τα πραγματικά συστήματα που υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα, όχι από τη δική μου τη δουλειά, αλλά από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε ε, το 2014, όπου κατεβλήθη προσπάθεια ανακεφαλαίωσης των συμπερασμάτων όλων των μελετών που υπάρχουν στον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική ε, που είναι πολύ δημοφιλής, όπου συγκεντρώνουμε αποτελέσματα από μελέτες, χιλιάδες μελετών για συγκεκριμένα θέματα και συγκρίνουμε ε, ζεύγη παρατηρήσεων ορίζουμε τον έλεγχο και συγκρίνουμε τον έλεγχο με την θεραπεία. Σε κάποιες μελέτες ε, ο έλεγχος είναι η παραδοσιακή βαθιά, το παραδοσιακό βαθύ όργωμα συγκρινόμενο με τις πρακτικές συντήρησης. Ε, υπάρχουν ε, μελέτες όπου εξετάζεται το μηδενικό όργωμα σε συνδυασμό με άλλα μέτρα και καταλήγουμε σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αυτά εδώ είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ε, δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα ως τα στοιχεία, αλλά αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι αυτή η τελεία δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά όσον αφορά την συγκομιδή ε, με βάση την συντηρητική και την παραδοσιακή γεωργία. Καμία διαφορά ε, στην απόδοση της ε, καλλιέργειας. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι κουκίδες που δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα, δεν προκύπτει μείωση της απόδοσης καλλιέργειας όταν χρησιμοποιείται η γεωργία συντήρησης. Έγιναν πάρα πολλές ε, μελέτες, ε, από 610 διαφορετικές μελέτες και διαπιστώθηκε, όπως σας είπα, ότι αν τελικά υπάρχει κάποια μείωση της απόδοσης, αυτή είναι ελάχιστη. Ε, υπήρξαν πειράματα όπου συμπεριλήφθηκε η αμυψή σπορά και η συγκράτηση του ύδατος η μείωση της απόδοσης ήταν κάπου μείον δύο, ελάχιστη δηλαδή. Η αμυψισφορά και η διαφοροποίηση των καλλιεργιών, αυτά ήταν τα βασικά πειράματα. Και στο τέλος βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη μείωση της καλλιέργειας ήταν όταν δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου το όργωμα και βλέπουμε τις ελάχιστες μειώσεις της, ε, των καλλιεργιών όταν οι τρεις πυλώνες εφαρμόστηκαν και οι τρεις από κοινού. Και βλέπουμε εδώ και πάλι τις ίδιες κουκίδες, όμως εδώ αναπαρίσταται και η κλιματική αλλαγή. Και βλέπουμε πάνω ότι όταν χρησιμοποιείται η γεωργία συντήρηση σε ξηρά κλίματα, ε, βλέπουμε ότι προκύπτουν ωφέλη, υψηλότερη απόδοση με την γεωργία συντήρησης από ότι όταν χρησιμοποιείται το παραδοσιακό όργωμα. Και αυτό ε, οφείλεται κυρίως στο ότι στα ξηρά αυτά κλίματα γίνεται καλύτερη συγκράτηση της ε, υγρασίας. Και κάτω βλέπετε σε πιο υγρά κλίματα, εκεί βλέπουμε κάποια μείωση της απόδοσης της καλλιέργειας. Άρα αυτό πρέπει κανείς να το έχει κατά νου, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, όπου με γεωργία συντήρησης μπορεί να υπάρχει μικρότερη απόδοση της καλλιέργειας. Εδώ μια εικόνα από το Newcastle. Βλέπετε στα δεξιά ε, το όργωμα, το παραδοσιακό και βλέπετε στην αρχή ε, της άνοιξης ε, και εδώ αριστερά είναι, δεν είναι τόσο έντονο το χρώμα ε, βλέπουμε λοιπόν αυτά τα πειράματα και έχουμε προβλήματα στα βόρεια κλίματα όπου έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενώ αλλού υπάρχει περισσότερη θερμότητα. Ε, είναι νομίζω κοινό αυτό στα βόρεια κλίματα. Βλέπουμε επίσης με την δομή του έδαφους, του εδάφους όταν υπάρχουν αμμόδιοι εδάφοι. Έχουμε, θέλουμε βιολογικά συστήματα, οι βιολογικές καλλιέργειες θέλουν να υιοθετήσουν τη γεωργία συντήρησης, διότι εξαρτώνται πάρα πολύ από το όργαμα. Θέλουν βεβαίως να ελέγξουν τα παράσιτα, τα ζυζάνια ε, και δεν έχουν αυτήν την επιλογή οι βιολογικοί καλλιεργητές. Θέλουν επίσης περιοδικά να οργώνουν ούτως ώστε να ενσωματώσουν και λιβάδια χωρίς να χρησιμοποιούν ζυζανιοκτώνα. Χρησιμοποιούν επίσης ε, κοπριές ε, οι οποίες είναι βιολογικές στο έδαφος και θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο ε, να υπάρξει ένα όργωμα στρατηγικό κατά καιρούς Επίσης θα πρέπει να καταστραφούν οι προστατευτικές καλλιέργειες, οι επικαλύψεις. Θα χρειαστούν λοιπόν ε, κάποιοι άλλοι τρόποι για να καταστραφούν. Αυτή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους βιολογικούς καραγητές, αλλά επίσης και τους συμβατικούς. Πρόκειται για ένα roller climper, ένα έλαστρο, και αν μπορούν κανείς στην κατάλληλη ε, στιγμή ε, να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα αυτό για την καλλιέργεια είναι η τεχνολογία που πρέπει να εξετάσουμε ούτως ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ε, για τα ζυζανιοκτώνα. Και έχουμε τελικά σχόλια θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα με, τις, ε, με τη γεωργία συντήρησης υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες οικοσυστήματος, αλλά υπάρχουν και προκλήσεις σε ορισμένα κλίματα, τα οποία είναι υγρά, τα οποία είναι κρύα κλίματα, και με συστήματα βιολογικά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα, θα πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογίες πιο κατάλληλες, ε, σπαρτικές μηχανές για γραμμική ε, σπορά ε, και αυτούς τους κυλίνδρους, τα έλαστρα, τα roller crimpers και επίσης καμιά φορά στο στρατηγικό όργωμα μπορεί να ενδείκνυται. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστούμε. Όπως σας είχα πει και προηγουμένως, μετά τους δύο πρώτους καλεσμένους, θα προβλέψουμε ένα χρόνο για ερωταπαντήσεις. Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο. Κύριος Αντές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ομιλίες σας. Ε, την πρώτη δεν την άκουσα ολόκληρη, δυστυχώς δεν ήρθα από την αρχή. 42 ε, εκτάρια έχουμε εμείς ε, στη δική μας την καλλιέργεια και προσπάθησα με την γεωργία στήριξη, αλλά δυστυχώς η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ αρνητική. και θέλω να σας πω ότι εντάξει δεν χρησιμοποιώ μεταξύ οπωσδήποτε μηχανές, όμως κάθε δύο χρόνια πρέπει να χρησιμοποιήσω μηχανική γεωργία. Αλλιώς θα μειωθεί κατά πολύ η απόδοση της ε, καλλιέργειάς μου. Μήπως ε, μπορείτε κι εσείς να τοποθετηθείτε λιγάκι από αυτού. Σε ποιον απευθύνετε εσείς την ερώτηση, σε ποιον την απευθύνετε. Ας μαζέψουμε πρώτα τις ερωτήσεις και μετά θα απαντήσουν οι προγνώμενες όλες μαζί τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, τις κυρίες ε, για τις παρουσιάσεις τους, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφορά τις εργασίες της Επιτροπής μας. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εμείς ε, Πρόσφατα ε, έχουμε εισάγει στην κοινή γεωργική πολιτική την αρχή του πρασινίσματος, ε, έτσι ώστε οι γεωργοί να χρησιμοποιούν πιο βιώσιμες ε, πρακτικές. Η ερώτηση που θέλω να κάνω, δεν ξέρω αν την έχετε κάνει εσείς, είναι κατά πόσον αυτές οι πρακτικές του πρασινίσματος που έχουμε εισαγάγει και υπάρχουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κάποια χρόνια, σχετικά με αυτές τις πρακτικές έχετε, έχετε κακή εμπειρία ή μήπως ε, τελικά ε, πρέπει κάπως να τροποποιηθούν αυτές οι αρχές έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη και αυτά στα οποία έχει καταλήξει η επιστήμη. Εμείς ε, την κάνουμε αυτή την ερώτηση γιατί το πρασίνισμα βεβαίως ήταν μια μεγάλη καινοτομία αλλά με το πρασίνισμα αυξήθηκαν κατά πολύ η γραφειοκρατία, τα προβλήματα των γεωργών. Εγώ λοιπόν θα ήθελα τελικά η προσπάθεια των γεωργών μας να επιβραβεύεται και θα ήθελα τη δική σας την άποψη από αυτού. Κυρία Σράιερ. Κυρία. Een beetje mis is eigenlijk de realiteit van vandaag. Wij beginnen niet opnieuw. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε. Στις ε, κάτω χώρες έχουμε την επόμενη χρονιά 500.000 αγελάδες που θα πρέπει να, μείνουν στις μονάδες. Δεν μπορεί κανείς από την μία μέρα στην άλλη να αλλάξει την κατάσταση. Μιλάμε για τις εξελίξεις στην Ήπεθρο. Είχαμε την πράσινη εβδομάδα. Είχαμε βεβαίως μεγάλα προβλήματα σχετικά με αυτό το οποίο πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα ε, να τα δούμε τα θέματα αυτά. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει την κατάσταση από τη μία μέρα στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ και τις ε, δύο πυρογνώμονες, ε, τις συγγήτριές μας σήμερα. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει προφανώς ε, και να καλλιεργούμε τη γη και όλοι συμφωνούν επίση ότι πρέπει να αποφεύγουμε τη διάβρωση του εδάφου. Το ερώτημα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ στο πλαίσιο του πρασινίσματο είναι το εξή. Μήπως ε, θα πρέπει τελικά να λέμε ότι ειδικά όταν πρόκειται για μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους, να καταλήγουμε σε περιφερειακά προγράμματα, όχι σε τοπικά ε, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλη σε έκταση και γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω και εγώ ε, κατά πόσον και εσείς συμφωνείτε ότι είναι καλύτερο να έχουμε περιφερειακά προγράμματα στην Ευρώπη ε, και όχι να πιστεύουμε ότι με τρία μέτρα πρασινίσματος σώσαμε τον κόσμο. Αυτό για μένα δεν αποδίδει. Δηλαδή δεν μπορούμε δυστυχώς με το πρασίνισμα να εφαρμόσουμε περιφερειακά προγράμματα και αυτό για μένα είναι πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Σουλαζό. Euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις ε, δύο μιλίες για το θέμα αυτό, το οποίο είναι σημαντικό. Αλλά μάλλον είναι ένας ισχυρισμό. Εγώ ε, ασχολούμαι με σιτηρά, είμαι γεωργός και είπατε ότι άμεση σπορά έχει ε, ωφέλη αλλά μείωση του κόστους. Όχι, δεν είναι παντού, διότι έχουμε ε, να κάνουμε, έχουμε μετά από 7 χρόνια, κάθε χρόνο έβλεπα ε, ε, ότι υπήρχε αλάτωση του εδάφους ε, και χρειάζεται να αγοραστεί υλικό που επιπλέον επιβαρύνει το κόστος και οι εργασίες αυτές στο έδαφος και επίσης βρωμίζει το έδαφος και θα πρέπει ότι αυτό το, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό από τεχνικής πλευράς, διότι είναι πολύ πιο περίπλοκο. Γι' αυτό σταμάτησα αυτήν την τεχνική και χρειάστηκε να επανεπενδύσω σε υλικό και όταν μιλάμε, δεν, μιλάμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μείωση του κόστους, είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει επιπλέον κόστος. Ο κύριος Φεράν. Euh, ναι, ε, τα φιλό, οι φιλόδοξοι στόχοι των κρατών μελών και η επιθυμία των Ευρωπαίων καταναλωτών δεν είναι κάτι το εφικτό ε, δυστυχώς ενώσω οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις ε, οι ευρωπαϊκές ε, σήμερα παίζουν για την επιβίωση τους λόγω της δραματικής κρίσης που παρατηρούμε σήμερα στην Ευρώπη. Και ακόμη και αν η στόχη αυτή είναι φιλόδοξη, ακόμη και αν είναι μια επιθυμία των Ευρωπαίων καταναλωτών, αυτές οι λύσεις δεν είναι εφικτές, δεν είναι πραγματοποιήσιμες. Ε, των, λόγω των δυσκολιών που γνωρίζουν οι γεωργοί με επιπλέον ε, της σύμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών της ΣΕΤΑ, βλέπουμε δυστυχώς ότι σήμερα δεν βλέπω πώς τέτοια μέτρα, τέτοιες προτάσεις θα μπορούν να έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ο κύριος Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις δύο μιλίες. Θα ήθελα να θέσω ε, για τα παρασιτοκτόνα μια ερώτηση. Ξέρετε ότι είχαμε μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απαγόρευση των ε, παρασιτοκτόνων, εκ των οποίων το μπιφοζάτα και ε, σύμφωνα με τη γνώμη σας στην επιστημονική μπορούμε να κάνουμε άνευ, διότι στην συμβατική γεωργία δεν μπορούμε διότι στα χρόνια όπου υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλή γρασία ε, και πολλές βροχές όπως είχαμε τον Ιούλιο στις χώρες μας και μετά έχουμε τα καπρίτσια του κλίματος δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς μη κοιτιοκτώνα και χωρίς παρασύτοκτώνα. Μπορούμε να σκεφτούμε μια γεωργία η οποία να είναι να απαλλαγεί από αυτού του είδους τα παρασιτοκτόνα στο μέλλον. Ο Άντριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για τις δύο ομιλίε και ευχαριστώ τον Μαρκ Καραμπέλα που μίλησε για τη γλυφοσάτη και αυτοί που έκαναν αυτή την επιλογή και στην Γαλλία. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ εν μέρη. Ε, βεβαίως, το Roundup για να γίνει αυτή η γεωργία, η γλυφοσάτη, το Roundup για να γίνει αυτή η γεωργία συντήρησης. Έχετε στοιχεία εξήγησης γιατί αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται ε, ε, ε, παγκοσμίω με συνέπεια και πολύ λίγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το κλίμα, είναι η γεωργία, είναι οι πρακτικές, έχετε αριθμούς, έχουμε στοιχεία. Και αυτό το ερώτημα είναι ουσιαστικό, διότι νομίζω ότι εγώ βλέπω πάρα πολλούς γεωργούς που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, που κάνουν μια εργασία πρόοδου, προσπαθούν ε, και από αγρονομικό ε, το, απόψεως και για να μπορέσουν να ξανακατακτήσουν εδάφη και είδωρ και πώς με την ερώτηση του κυρίου Ντεκάστρο μπορούμε να κάνουμε στην ΚΑΠ να βελτιώσουμε το θέμα και ίσως να απλουστεύσουμε με αγρονομική προσέγγιση ε, και να βγούμε από το, το, το διοικητικό, ε, ποιοτικό, αγρονομικό θέμα ε, προς όφελος των γεωργών. Η κυρία Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις δύο καλεσμένες μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Μήπως θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο στο θέμα του αντικτύπου αυτής της γεωργίας συντήρησης ε, στη δέσμευση του άνθρακα. Και δεύτερον, η αγροοικολογία είναι λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα διαφύλαξης του εδάφους από ότι η γεωργία συντήρησης. Ευχαριστώ κυρία Νόιχλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον που συζητάμε για το έδαφος, γιατί κατά κανόνα συζητάμε εδώ για κονδύλια ενισχύσεων, ε, για ε, λοιπάσματα, αλλά εγώ πιστεύω στη Γεωργία το σημαντικότερο είναι το έδαφος. και αν θέλουμε πραγματικά ένα υγιές έδαφος πρέπει να συζητήσουμε επ' αυτού έγινε λόγος για το Roundup. Ε, υπάρχουν ε, στη Γερμανία πάρα πολλές ομάδες που ασχολούνται ακριβώς με αυτή τη μορφή επεξεργασίας ε, του εδάφους. Ξέρετε, μπορεί κανείς να μειώσει την πίεση στο έδαφος και με τον τρόπο αυτό να είναι δυνατόν να απορροφάτε καλύτερα το νερό στο έδαφος. Θέλω να μα μιλήσετε λιγάκι από αυτού για την απορροφητικότητα του εδάφους. Αυτό είναι το ένα που με ενδιαφέρει. Και το δεύτερο είναι στι ε, στις βιολογικές ε, Γιατί θεωρείτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή η μορφή γεωργία Εδώ κατ' ουσίαν ε, πρόκειται για επικάλυψη απόψεων και μεθόδων. Γιατί λοιπόν στον βιολογικό τομέα η, γεωργία, η, συντηρητική γεωργία αυτή για την οποία συζητάμε σήμερα, γιατί αυτή δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Γιατί δεν τη συζητάνε, δεν την προβάλλουν τόσο πολύ τη γεωργία συντήρησης. Ναι, ε, ευχαριστώ για τις ομιλίες. Ανεξάρτητα από τα θέματα απόδοσης και ε, για το τι περιλαμβάνεται. Αυτό που με ενδιαφέρεται είναι το θέμα της διάβρωσης των εδαφών ε, που ε, έχει επιπτώσεις πάνω στο υδραυλικό δίκτυο και πάνω στην Πανίδα και στη Χλωρίδα. Το διαρωτώ με εάν ποια είναι η καλύτερη πρακτική, η κάλυψη, η φυτική που προτείνεται ή ε, ορισμένες φυτεύσεις ε, που να μπορούν ε, να μας κάνουν να αποφύγουμε τη διάβρωση. Είδαμε πώς αλλάζει η γεωργία, πώς από επεκτατική γίνεται εντατική και κρυζώνοντας ορισμένα, ορισμένα φυτά έχουμε επιπλοκές όσον αφορά το είδωρο. Σας ευχαριστώ κύριε Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι δύο ομιλίες. Ε, μαθαίνουμε κάτι καινούριο κάθε μέρα όταν ερχόμαστε εδώ. Βεβαίως είναι όπως για την βιολογική ε, γεωργία. Φαίνεται βεβαίως, όπως είπε κι άλλος ομιλητής, αν υπάρχει ε, τρόπος να περάσουμε σε αυτό, δεν ξέρω ε, είχαμε ε, στο γραφείο μου πάρα πολλές εντελεχείς ε, συζητήσεις και ένας από τους οικολόγους που μίλησε για το ίδιο θέμα και μιλούν ακόμα και συζητούν για την χλυφοσάτη. Και νομίζω πόσο εφικτό είναι να μπορεί κανείς γεώμηλα ή να έχει άλλες καλλιέργειες χωρίς να χρησιμοποιείται. Νομίζω θα ήταν καλό αν ε, ήμασταν ε, χιλιάδες μίλια μακριά από αυτό που ακούμε και θα θέλαμε, ε, διαρωτώ με επίσης, για αυτό που είπατε για το ρόλο της βελτίωσης του εδάφους του αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο και, και στο TTIP, στο Mercosur γίνεται λόγος γι' αυτό. Μήπως ενδιαφέρεστε για αυτές τις συμφωνίες. Τι θα γίνει με αυτές τις συμφωνίες. Θα καταστήσουν πιο πιθανό ή λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ κύριο Σάγνιο. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ προσπαθήσω στον Ηνωμένο Βασίλειο να ζητήσω φαινόμενα διάβρωσης, θα δω ότι είναι, οφείλονται σε τρεις ε, αιτίε. Καταρχήν ε, έχουμε όσο πιο βαθύ είναι το όργαν, όργωμα, πιο βαθίε βαθιές είναι οι που δημιουργούνται κατά το τόσο πιο εύκολα διαβρώνεται. Τι κάνουμε όμως εδώ στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ενθαρρύνουμε για ακόμη μεγαλύτερο ψεκασμό ε, για να χρησιμοποιούνται ζενιοκτώνα και, να, ε, και φυτοφάρμακα για να εξοντωθούν μερικά ζωήφια. Τώρα όλο και περισσότερο γίνονται ψεκασμοί ε, ή χρησιμοποιούνται κάποια ρουρέ για να φάνε αυτά τα ζωήφια και τα αυλάκια γίνονται ακόμη πιο βαθιά με αποτέλεσμα η διάβρωση να είναι ακόμη πιο έντονη. Επίσης, αλλού που βλέπω διάβρωση στο Ενωβέρα Βασίλειο ε, καταρχήν, όταν έχουμε υγρό καιρό, βροχοπτώσει τον Εύρη για παράδειγμα, και θέλουμε καλλιέργειες ε, ε, βολβών και ριζών, όταν γίνεται εσοδεία τέτοιων ριζών σε βροχερούς καιρούς υπάρχει πρόβλημα. Και το καταλαβαίνω αυτό που έχουμε τα γεώμηλα, το πρόβλημα Ιρλανδί. Επίσης, τα ζώα δεν μπορούμε τις, τις Άγια Ελλάδες μας τις κρατάμε ή τα, τα, τους χείρους ε, στους ε, σταύρους και στα χειροστάσια, είναι, είναι λογικό να θέλουν να βγαίνουν έξω, να βόσκουν ελεύθερα. Οπότε με αυτά τα τρία φαινόμενα έχουμε διάβρωση. Τι να κάνουμε, να κρατάμε τους χείρους στα χειροστάσια ή να τα αφήνουμε έξω να έχουμε έτσι χείρους ελευθέρας βοσκής και άλλα να υποφέρει το έδαφος από διάβρωση. Επίσης, ε, το το να συνδέεται το διοξείδιο του άνθρακα και τη μείωση της ε, κατανάλωσης ενέργειας. Εντάξει, καλή μείωση η κατανάλωση ενέργειας. Τώρα μιλάτε όμως για ε, διοξείδιο του άνθρακα. Μα το διοξείδιο του άνθρακα είναι καλό για τις καλλιέργειες. Όσο περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει, τόσο πιο μεγάλη είναι απόδοση, τόσο πιο γρήγορα μεγαλώνουν τα φυτά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συνδυάζεται το, ε, την, τη μείωση του κόστους και την... Ε, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό είναι απολύτω ασφαλμένο. Επίσης, αν αφήσουμε για, σε αγρανάπαυση λίγο τα εδάφη, θα αναδιαρθρωθούν από μόνα τους. Οπότε δεν χρειάζεται να τα ε, βοηθάμε εμείς, αρκεί να τα αφήσουμε λίγο ήσυχα. Επίσης, ε, τελικά με τη μηδενική άρρωση δεν είναι σίγουρη ότι η υποδοτικότητα θα είναι η αναμενόμενη. Μερικές φορές είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Και είπατε ότι ήταν τεράστιο το κόστος που γλίτωσαν οι γεωργοί. Είναι όντως ε, μεγάλη αυτή η οικονομία που γίνεται. Γιατί εμείς είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα με πραγματικές εξοικονομήσεις. Ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τώρα, ε, για της, για τη ρηχή, τη μηδενική άρρωση έχει νόημα για ορισμένε καλλιέργειες, όχι για τις ρίζες. Τώρα για την κλειφωσάτη. αν θέλετε να καταργήσετε, να απαγορεύσετε την γλυφοσάτη, ξεχάσετε τη μηδενική άρρωση στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε και το ένα και το άλλο. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το πώς αυτά τα συστήματα επηρεάζουν τη διαχείριση των υδάτων στις αρδεύσεις. Έχετε πέντε λεπτά η καθεμία παρακαλώ. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ τις πολυάριθμες ερωτήσεις που μας υποβάλλατε. Δεν ξέρω αν μου διαφύγει καμία να με συμπαθάτε. Είναι σίγουρο ότι οι γεωργίες συντήρησης δεν είναι πανάκια. Δεν πρόκειται να έχουμε καμιά θαυματουργή λύση και από το πρώτο έτος να έχουμε αμέσως ε, μερικά ή όλα από τα ωφέλη που σας περιέγραψα. Για παράδειγμα, η απορροές, ε, η απώλεια ύδατος και η διάβρωση, όντως ε, θα φανεί από την αρχή, αλλά η γονιμότητα δεν θα φανεί αμέσως βραχυπρόθεσμα, χρειάζεται χρόνος για να αποκατασταθεί, να αυξηθεί η γονιμότητα του εδάφους. Σε ό,τι αφορά τη γλυφοσάτη που ανέφεραν κάποιοι ευρωβουλευτές, ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η συμβατική γεωργία και όχι η γεωργία συντήρησης χρησιμοποιούν τη γλυφοσάτη. Εμείς δεν έχουμε ούτε 4 εκατομμύρια εκτάρια γεωργία συντήρησης, ε. οπότε είναι περιθωριακή χρήση γλυφοσάτης από τη γεωργία συντήρησης. Και μάλιστα μπορούμε να έχουμε και γεωργία συντήρησης ε, και να μην χρειαζόμαστε αυτό το ζυζανιοκτόνο, τη γλυφοσάτη. Θα μπορούσαμε ίσως να το αντικαταστήσουμε με ένα πιο επιλεκτικό ζυζανιοκτόνο και όχι τη γλυφοσάτη που είναι ο και τα καταστρέφει όλα. Η κυρία Κούπερ μας ανέφερε κάποιες μηχανές, κάποια μηχανήματα που υπάρχουν και μπορούν να κάνουν το ξεβοτάρισμα μηχανικά με αυτούς τους τροβίλους που έχουν και τα ελάσματα. Σε ό,τι αφορά το έδαφος, ο κύριος Άλμπερτ Ντες έθεσε μία ερώτηση. Θα ήθελα να του πω ότι μακροπρόθεσμα βλέπουμε πλέον ε, αλλά πρέπει να περιμένουμε για άλλα τα πλεονεκτήματα είναι πιο βραχυπρόθεσμα. Σε ό,τι αφορά το όργωμα, την άρρωση, τα εδάφη είναι διαφορετικά. Υπάρχουν εδάφη που κάνουν ένα είδος αυτοάρρωση από μόνα τους. Αν όμως θέλουμε εμείς να οργώσουμε, δηλαδή να μακιγιάρουμε κατά κάποιο τρόπο το έδαφος, θα πρέπει να κάνουμε ένα ξεβοτάνισμα, να ξεριζώσουμε κάποια ζυζάνια, γιατί φυσικά δεν θέλει ο Γιώργος να βλέπει ζυζάνια στο χωράφι του και με το όργωμα και αυτό κάνουμε. Αλλά το έδαφος από μόνο του δεν χρειάζεται άρρωση μηχανική. Σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα τώρα. Το ανέφεραν ο κύριος Κάστρο και κάποιοι άλλοι. Όπως είπα και προηγουμένως, ούτε μόνο με τον Greening και τις άμεσες πληρωμές της ΚΑΠ και δεν ξέρω βέβαια αν κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τη γραφειοκρατία, γιατί στόχος είναι η απλοποίηση, η απλούστευση της γραφειοκρατίας. Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες ε, και επιλογές στον ε, Γεωργό. Όχι μόνο άμυψη σπορά ε, ή τα μέτρα του greening για να μπορέσει να διαφυλάξει την ποιότητα του εδάφους του γιατί η γεωργία συντήρησης προποθέτει κάποιες τεχνολογικές ε, εξελίξεις και τεχνολογική πρόοδο και είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ε, επικουρικά τη συντηρητική γεωργία με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Γιατί όλοι οι γεωργοί ε, πρέπει να εκπαιδευτούμε στις νέες πρακτικές. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε ένα σύστημα διαχείριση του εδάφου εν μία νυχτή, χωρί προηγουμένω να μην έχουμε επιμορφωθεί για τη νέα πρακτική. Οπότε στο δεύτερο πυλώνα τη ΠΑΚ, τη ΚΑΠ, συγγνώμη, και σε περιφερειακό επίπεδο, όπω αναφέρθηκε, θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνικές και να προσαρμόσουμε τις νέες τεχνικές γεωργία συντήρησης στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μέσω του δεύτερου πυλώνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βελτίωση της διείσδυσης του ύδατος στο έδαφος, χάρη στη γεωργία συντήρησης, υπάρχει βελτίωση της ε, διείσδυσης του ύδατος και αποφεύγεται η συμπίκνωση και ακριβώς επειδή δεν έχουμε συνεχώς ε, μηχανές που να οργώνουν, το έδαφος ε, δεν, έχει, δεν υφίσταται τέτοια συμπίκνωση, οπότε και το νερό διεισδύει καλύτερα. χάρη στη μία άρρωση, η διείσδυση του νερού μέσω και μακροπρόθεσμα θα βελτιωθεί στη γεωργία συντήρηση. Έχουμε πολλές μελέτες, όχι μόνο στην Ισπανία και σε άλλες χώρες, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες ε, τρίτες χώρες γίνονται μελέτες ε, που το τεκμηριώνουν. Ο κύριος Ταραβέλα μίλησε για τη διάβρωση και ρώτησε πώς μπορούμε να προλάβουμε τη διάβρωση. Φάνηκε και από τις φωτογραφίες που σας έδειξα ότι και σε μονοετής αλλά και σε πολιετής καλλιέργειες ε, αποφεύγουμε την διάβρωση αν κρατάμε καλυμμένο το έδαφος. Μερικές χώρες χρησιμοποιούν τις προστατευτικές καλλιέργειες, τις αντιδιαβρωτικές, τις καλλιέργειες βλαστικής κάλυψης ή χρησιμοποιούν τα υπολείμματα προηγούμενων καλλιεργειών. Η γεωργία συντήρησης δεν ξεκινά με τη σπορά αλλά με την ε, συγκομιδή της προηγούμενης καλλιέργειας. Για παράδειγμα, μαζεύουμε το σιτάρι και ταυτόχρονα συλλέγουμε όλα τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας. Έτσι κρατάμε καλυμμένο το έδαφος και για τις ε, μεταγενέστερες πόρες. Και να ολοκληρώσω ε, μιλώντας για τα γιόμιλα που μας ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που γίνεται κυρίως στη Γαλλία και εκεί έχουμε πατατοκαλλιεργητές στη Βόρεια Γαλλία, κοντά στο Καλέ, που χάρη στις ανεψισπορές που εφαρμόζουν, 6-7 διαφορετικές εναλλακτικέ καλλιέργειες, έχουν πολύ καλές αποδόσεις στις εσοδίες ε, πατάτας, χάρη στις τεχνικές της γεωργίας συντήρησης.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 Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτήτικα, δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Αλλά και η συνάδελφός μου απάντησε. Υπάρχει κάτι που μου έχει κάτσει στο μυαλό. Το ένα είναι τα οικονομικής φύσεως θέματα, τα οποία προέκυψαν σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, νομίζω ότι δεν τα εξηγήσαμε καλά τα οικονομικά. Αυτό που ε, είπε, αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, ήταν ότι όλα αυτά κοστίζουν περισσότερο. Ε, πολλοί είπαν ότι όλα αυτά είναι δαπανηρά να εφαρμοστούν στην Γαλλία. Αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί ο κύριος Αγγνιού έχει δίκιο που είπε ότι όσοι γεωργοί στην ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν γεωργία συντήρησης, το κάνουν για να εξοικονομήσουν ε, κόστος ενέργειας και προσωπικό και επίσης το κέρδος είναι υψηλότερο. Τουλάχιστον αυτό ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύει στη Γαλλία. Το άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, Βεβαίω, ε, οι ε, γεωργοί δεν θα καταλήξουν σε κάτι αν δεν υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Κατά τα άλλα, έγιναν και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το γιατί δεν χρησιμοποιείται η ε, γεωργία συντήρησης στις οργανικές, στις βιολογικές καλλιέργειες. Νομίζω ότι μίλησα γι' αυτό στην ομιλία μου. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις ε, βιολογικές καλλιέργειες. Ε, έχουμε την χρησιμοποίηση των ζανιοκτώνων για τα παράσιτα ε, και οι βιοκαλλιεργητές ε, ε, οποτεδήποτε δεν οργώνουν βεβαίως και βλέπουν ότι εμφανίζονται περισσότερα παραστοκτόνα. Άρα δηλαδή οι γεωργοί οποτεδήποτε περνάνε στην καλλιέργεια την, με τη συντήρηση προφανώς και προκύπτουν περισσότερα παρασιτοκτόνο. Αλλά αυτό ε, δεν σημαίνει απαραίτητα μικρότερη απόδυση. Ε, ίσως λοιπόν θα πρέπει ε, στο πλαίσιο της συντηρητικής γεωργίας, της γεωργίας συντήρησης, να υπάρχει και κατά κάποιο όργαμα. Στα, στις βιοκαλλιέργειες χρησιμοποιείται το όργωμα για να αντιμετωπιστούν τα ζυζενιοκτώνα, τα οποία ενδεχομένως έχουν προκύψει. Όπως σας είπα λοιπόν, ε, η γεωργία συντήρησης θα πρέπει να προσαρμοστεί λιγάκι. Ο κύριος Φλάναγκαν είπε ότι ε, θα πρέπει κανείς να δει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και το όργωμα ε, στην καλλιέργεια στην υγειοργία συντήρησης. Όπως σας είπα θα πρέπει να υπάρχουν προσαρμογές. Επίσης μιλήσατε για την βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Ε, δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολύ ε, μεγάλη εμπειρία από αυτού. Πάρα πολλοί έκαναν μια ερώτηση ε, κατά πόσον μπορεί να αντικατασταθεί η γλυφοσάτη. Προφανώς και μπορεί να αντικατασταθεί και να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα, ε, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Νομίζω ότι υπήρξε και κάτι άλλο που ήθελα να απαντήσω. Αυτά, μάλλον αυτά. Νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ για τις ε, πάρα πολύ καλές ερωτήσεις, ε, γιατί από ό,τι φανείται τελικά οι καλές αυτές ερωτήσεις έδειξαν ότι μας προσέξατε, μας παρακολουθήσατε στις ομιλίες μας. Σας ευχαριστούμε. Εννοείται. Επιτροπή Γεωργίας είμαστε. Αλλήμωνα δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά τα θέματα. Παρακαλώ τώρα την επόμενη μας εμπειρογνώμονα να έρθει στο βήμα. θα λάβετε θέση, παρακαλώ. E, e, έχουμε την κυρία Μότσα. Ε, έχουμε και την κυρία ε, ε, η Αγγλία από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητή έχει ασχοληθεί με πολλά θέματα ευημερία των ζώνων ευζοία, καλής μεταχείρισης, αλλά και για πολλά και διάφορα θέματα. Την καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση και χαιρόμαστε πολύ γιατί θυμόμαστε τη φοβερή συνεισφορά της ε, στα ζητήματα της Γεωργίας από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ε, Έχουμε λοιπόν δύο ακόμη εμπειρογνώμονες, ε, όπως σας είπα και προηγουμένως, την κυρία Εύα Ρεμότσα. που είναι ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Παύλο Δολαβίτε της Σεβίλης και κατόπιν τον κύριο Έκτορ Μολίνα Φάμπρα, καθηγητή γαστρονομίας. Ε, πρώτα κυρία Τόρε Μότσα, γιατί ακολουθούμε τη σειρά του προγράμματος. Muchas Σας ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω ένα πρόβλημα με την πτήση μου. Σε 20 λεπτά πρέπει οπωσδήποτε να φύγω. Γι' αυτό και θα κάνω πολύ σύντομη την παρέμβασή μου, ώστε να μείνει λίγο χρόνο για να υποβάλλετε τι ερωτήσει. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά υπήρξε μια αλλαγή δυστυχώ. Δεν καταφέραμε να συντονιστούμε καλά και πρέπει να φύγω για την πτήση μου σε 20 λεπτά. Όπω σα είπα, εγώ προέρχομαι από την αγροοικολογία, από τον κόσμο τη βιολογική γεωργία και θα ήθελα να διατρανώσω την αμέριστη υποστήριξή μου ε, εκ μέρου τη βιολογική γεωργία, του κόσμου τη βιολογική γεωργία, την αμέριστη υποστήριξή μα στην γεωργία συντήρηση. Παρόλο που έχω για κάποιε κριτικέ και πιστεύω ότι επιδέχεται βελτίωση αυτό το θέμα. Πάντω, ε, σίγουρα αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση τη γεωργία συντήρηση. Στη συνέχεια θα σα ε, εξηγήσω γιατί η βιολογική γεωργία μπορεί να δώσει κάποιες βασικούς άξονες και βασικές κατευθύνσεις και να σας πω ότι βρισκόμαστε συνεχώς ε, σε μια μεταβατική φάση, γιατί διαπιστώνουμε ότι η γεωργία μας πια δεν είναι βιώσιμη. Και αυτό το αναγνωρίζουμε πια σχεδόν όλοι. Αντιμετωπίζουμε σοβαρότατες ε, προκλήσεις όπως τις κλιματικές αλλαγές, την πείνα, την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, την ε, εναλλαγή των γενεών στη γεωργία γιατί εδώ και χρόνια έχουμε ένα γυράσκοντα αγροτικό πληθυσμό και δεν υπάρχει σκητάλη, να δίνεται σκητάλη από τη μία γενεά στην άλλη, κάτι που δεν πρόβλημα που δεν έχουν ούτε στη Λατινική Αμερική ούτε στην Ινδία. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ε, την επισητιστική μας ασφάλεια από τη Γεωργία. Έχουμε μια συστημική λοιπόν προσέγγιση που χρειαζόμαστε και θα πρέπει να δούμε και το θέμα της βιωσιμότητας, γιατί έχουμε πολλά θέματα που δεν αφορούν μόνο την καλλιέργεια, αλλά και τη γεωργία ως βασικό παράγοντα επισητισμού. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτή την παραγωγή τροφίμων, γιατί αυτό το στόχο γεωργία, την παραγωγή τροφίμων. Να κάνουμε μια σύντομη σύγκριση μεταξύ γεωργίας συντήρησης και βιολογικής γεωργίας, αγροοικολογικής μάλιστα. Ε, επίπτωση τη γεωργία συντήρηση βρίσκεται στα εδάφη, ενώ η ε, ε, αγροεκολογία, έχει χρησιμοποιεί το έδαφο ε, ω βάση τη παραγωγή, αλλά λαμβάνει υπόψη και το είδωρ και τη βιοπικιλότητα, οπότε ο δικό μα αντίκτυπο δεν περιορίζεται μόνο στο έδαφο. γιατί ναι, βέβαια δεν χρησιμοποιούμε λιπάσματα και δεν μολύνουμε του υδροφόρους ορίζοντες, αλλά ο αντίκτυπό μα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Επίση, στην κλίμακα μεγέθου η γεωργία συντήρηση περιορίζεται στο αγροτεμάχιο. Ενώ εμείς στην αγροοικολογία μιλούμε για τοπία, για γεωργικά τοπία, για ευρύτερα εδάφη. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την προσέγγιση μας, να μην περιοριστούμε στο αγροτεμάχιο, αλλά στο, στα ευρύτερα εδάφη, στα τοπία, που θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση γιατί είναι περίπλοκη η γεωργία. Επίσης, μιλούμε για καλλιέργειες αλλά και για μυψισπορές. Εναλλαγή καλλιεργειών απαραίτητο, απαραίτητη προϋπόθεση για να αναχαιτήσουμε τη διάβρωση. Έχουμε το πρόβλημα με τα ζυζάνια, το αναγνωρίζουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και στο μέλλον να βρούμε κάποιες λύσεις γιατί τα ζυζάνια τρώνε τις καλλιέργειες παρόλο που υπάρχουν τεχνικές και στρατηγικές να μειώσουμε κάπως την επέλαση των ζυζανίων. Γεωργικές ισουραές. Μειώνονται οι ισουραές στην γεωργία συντήρηση, ε, χρησιμοποιούνται καλύτερα και γίνεται καλύτερη εξοπλίση των χημικών. Εμείς θέλουμε να μην είναι τοξικά αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Βέβαια, δεν διεκδικούμε βιολογική γεωργία παντού και παγκοσμίω, αλλά θα πρέπει ε, να θεωρήσουμε τη γεωργία συντήρησης ως πρώτο στάδιο για να ε, μεταβούμε σταδιακά προς μια γεωργία χωρίς τοξικά προϊόντα. Φυσικά θα γίνει εν μία νυχτή. Επίσης, ποια είναι τα ωφέλη, μείωση της ε, διάβρωσης, ε, αύξηση της ε, υγρασίας του εδάφους, που είναι σημαντικό ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου, και επίσης η οργανική ύλη αποτελεί τη βάση της αναπαραγωγής του συστήματος, γιατί έτσι θα μπορέσει το σύστημα παραγωγής να διαφυλαχθεί και όσο πιο μεγάλη αυτονομία έχει το σύστημα στη διατήρησή του, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα θα αποκτήσει και μεγαλύτερη ικανότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ε, της βιωσιμότητας και των κλιματικών αλλαγών. Εμείς ε, μειώνουμε και την ε, μόλυση του εδάφους, αλλά και τη μόλυση των υδάτων. Συνεχίζουμε τις συγκρίσεις. Ποιος είναι ο ρόλος της φύσης, του πλαισίου, του συστήματος στο οποίο κινούμαστε, στην ε, γεωργία Συντηρής είναι πιο παθητική η στάση. Είναι ένας άνθρωπος, ένας γεωργός που δρά στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, αλλά η γεωργία είναι κάτι πολύ ευρύτερο, είναι ένα ζωντανό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβει και τη φύση που έχει ρυθμιστικό ρόλο και θα πρέπει να τον αναβαθμίσουμε και να τον αξιοποιήσουμε, να μην επαναπαυτούμε στις δράσεις μας θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτέ τι ρυθμιστικέ δραστηριότητε, να ερευνήσουμε σε αυτέ και να τι ενισχύσουμε ώστε να αυξήσουμε την παραγωγή των τροφίμων με τεχνικέ όμω που θα είναι βιώσιμε. Η υπηρεσία των οικοσυστημάτων και η δέσμευση του άνθρακα. Γίνεται αυτό στη Γεωργία Συντήρηση και μάλιστα πρόσφατε μελέτε, Ρώσιν και όλα, μα λένε ότι επιπλέον στην βιολογική γεωργία, χάρη στην συμπερίληψη οργανικών υλικών, που τα προσθέτουμε, όχι απλώς αξιοποιούμε αυτά που υπάρχουν, γιατί η γονιμότητα του εδάφους είναι κλειδί και σε αυτή την οργανική ύλη γίνεται η δέσμευση του άνθρακα. Εμείς απαιτούμε να ισχύσει κάτι τέτοιο, όχι να διατηρήσουμε τη γονιμότητα, αλλά να την ενισχύσουμε κιόλα, γιατί αυτό κατά τη γνώμη μας είναι κλειδί της ζωής του εδάφους και κλειδί για την παραγωγή τροφίμων. Επίσης γνώσεις, όχι μόνο τεχνικές που είναι χρήσιμες, αλλά θέλουμε και ε, τοπικές γνώσεις για το κλίμα, τις περιφέρειες, Θέλουμε ε, την τοπική γνώση και των γεωργών που έχουν εμπειρικές γνώσεις και συμβάλλουν ε, στην συγκέντρωση περισσότερων γνώσεων και την ανέβρεση λύσεων στο βιοφυσικό και πολιτιστικό αυτό περιβάλλον. Επίσης, ε, εντατικοποίηση, που είναι μια λέξη της μόδας. Θέλουμε αύξηση της παραγωγής για να καταπολεμήσουμε την πείνα. Θέλουμε όμως μια βιώσιμη γεωργία. Δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη εντατικοποίηση όταν στηριζόμαστε σε μια επανάληψη του μέχρι τώρα μοντέλου που απέδειξε ότι δεν είναι βιώσιμο. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουμε στην αγροοικολογία ε, να αυξάνουμε τις γνώσεις μας για τον ρυθμιστικό ρόλο της φύσης και να επενδύσουμε στην καινοτομία, στα drones ε, και οι γεωργίες συντήρηση δεν είναι ασύμβατη με την αγροοικολογία. Επαναλαμβάνω, είναι συμπληρωματικέ. Και τώρα τι μοντέλο χρειαζόμαστε. Ε, εμείς θέλουμε ένα συστημικό μοντέλο, περιεκτικό, ολιστικό, για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες αυτές προκλήσεις και τις αλλαγές. Το αγροτεμάχιο είναι ένα τμήμα του κόσμου, είναι μια ψηφίδα του παζλ. Αν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας και να αντιμετωπίσουμε τη γεωργία ως μια ευρύτερη υπηρεσία και ως ένα πολυδιάστατο χώρο, πλουραλιστικό, πολυδιάστατο, πολυσχηδή. Γι' αυτό και θα πρέπει ε, να υιοθετήσουμε μια τέτοια πολυσχηδή προσέγγιση. Δεν αρκεί μια οριζόντια προσέγγιση για να υλοποιήσουμε το στόχο μας, γιατί θα φτάσουμε γρήγορα στα ωριά του. Έδειξαν οι μελέτες ότι η βιολογική γεωργία δεσμεύει πολύ περισσότερο άνθρακα στα πρώτα 30 εκατοστά του εδάφους. Χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, γιατί η αυτονομία είναι από τα βασικά κλειδιά της ε, βιολογικής γεωργίας και εξαρτάται όλο και λιγότερο από τις γεωργικές εισρωές. Οι ε, εισρωές προέρχονται από το τοπικό πλαίσιο για να περιορίζονται τα κόστη της μεταφοράς ενέργειας. Επίσης έχουν μεγαλύτερη ενθεκτικότητα στην ξηρασία από την γεωργία συντήρησης. Γιατί ακριβώς προσθέτουμε γεωργική ύλη στο έδαφος για την παραγωγικότητα. Εκεί κάπως υστερούμε, το δείχνουν και οι μελέτες και το αναγνωρίζουμε και εμείς. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Δεν θα σας πουλάμε εδώ λαγούς με πετραχίλια, αλλά έχουμε το ίδιο επίπεδο παραγωγικότητας με την συμβατική γεωργία αυτός είναι, αυτός είναι ο στόχος. Θα πρέπει όμως να αξιοποιήσουμε αυτή τη συστημική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που είναι πολυδιάστατες. Για παράδειγμα, η αλλαγή της διατροφής είναι ένας άλλος τρόπος, γιατί ε, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο κρέας. Και από τη γεωργία θα έρθει ένα τμήμα της λύσης, αλλά θα πρέπει να να δούμε και άλλα θέματα και εντός του αγροεπιστηστικού κλάδου και εκτός. Επίσης να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων. Γιατί δεν θα πρέπει να παράγουμε τρόφιμα που θα καταλήγουν στα σκουπίδια. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση των τροφίμων και να αποφευθεί η κατασπατάληση τροφίμων. Και η εντατικοποίηση που ζητάμε, αν περιορίσουμε τη σπατάλη, θα περιοριστεί και αυτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν παραγωγικά συστήματα που να είναι σχεδιασμένα σε μεγαλύτερη κλίμακα από την παραγωγική μονάδα και χρειαζόμαστε και συστήματα που να μα το επιτρέπουν. Και ευτυχώ η ΚΑΠ κάνει αυτό το πρώτο βήμα τη συμπερίληψη και άλλων πτυχών στη διαχείριση. Όπω έχουμε την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση Καινοτομία. Ε, χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, ε, θέλουμε και κατακόρυφη και οριζόντια ολοκλήρωση δεν θέλουμε μία μονοσήμαντη πορεία. Είναι πολλές οι προκλήσεις και η προσέγγιση θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη. Επίσης, ε, πολλοί γεωργοί έχουν κάνει τις επιλογές τους και εφαρμόζουν κάποιες καινοτόμες τεχνικές. Βέβαια, οι αλλαγές δεν θα γίνουν ε, από τη μία μέρα στην άλλη, το 2020, το 2030. Έχουμε ορίζοντα το 2050. Θα πρέπει να καλύψουμε τις ελλείψει που έχουμε στην έρευνα και να συμπληρώσουμε τις ελλείψεις που έχουμε και στα τεχνικά θέματα και που χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και καλύπτονται. Σας ευχαριστώ. Είπατε ότι έχετε πολύ λίγο χρόνο, γι' αυτό και θα δώσω τώρα την ευκαιρία στους συναδέλφους να σας θέσουν ερωτήσεις, μια και πρέπει να φύγετε σε λίγο. Η κυρία Αγγιλέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, καταλαβαίνω ότι ε, για σας, ε, τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας, η γεωργία συντήρηση είναι μια πρώτη φάση μόνο, το πρώτο βήμα. Αλλά δεν κατάλαβα αν αυτή η συμβίωση μεταξύ της γεωργίας συντήρησης και της οικολογικής γεωργίας ή της βιολογικής γεωργίας ε, είναι απόλυτα σωστή. Γιατί στην αρχή είπε ότι γίνεται, μετά μου δημιουργήσει κάποιε αμφιβολίε για αυτή τη συμβίωση. Ποια είναι αυτή η πρώτη φάση, κατά τη γνώμη σου. Σίγουρα θέλουμε το έδαφο μας να είναι ζωντανό, να έχει οργανική ύλη. Και όλες ε, οι τεχνικές της ε, γεωργία συντήρηση έχουν στόχο αυτή τη διαφύλαξη τη οργανική ύλη στο έδαφο. Θέλουμε λοιπόν ένα ζωντανό έδαφο. Από τη στιγμή που έχουμε ζωντανό έδαφο, θέλουμε να αυξηθεί αυτή η ζωτικότητα, να μειώσουμε δηλαδή τη χρήση τοξικών προϊόντων ή κάποιων συστατικών που μπορεί να περιορίσουν την πανίδα του εδάφου, να σκοτώσουν την πανίδα του εδάφου. Ξέρουμε ότι απαγορεύτηκαν δύο ζυζανιοκτώνα γιατί σκοτώνουν τι μέλισσε. Ε, Πολλέ φορέ η μικροπανίδα του εδάφου ε, περιορίζεται εξαιτία τη έκθεση σε χημικού και τοξικού παράγοντε. Επίση, θεωρώ ότι η γεωργία συντήρηση είναι ο σύμμαχο τη βιολογική γεωργία. Θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση ε, χημικών ουσιών. Αυτή είναι η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση είναι η συμπερίληψη του, της περιοχής στην, ε, στον αγροεπιστητικό σχεδιασμό. Επίσης, ε, να έχουμε μια αυτονομία των γεωρικών ισρών και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την κομποστοποίηση, ώστε τα υπολείμματα των καλλιεργιών να χρησιμοποιηθούν, να αυξηθεί η ζωτικότητα του εδάφους, να αυξηθεί η οργανική ύλη και έτσι θα μειώσουμε τον αντίκτυπο ή το κόστος της συμβατικής γεωρικής παραγωγής. Αυτά θα γίνουν φυσικά αργά, με αργά αλλά σταθερά βήματα. Ευχαριστώ κυρία Σλάιερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πραγματικά αυτά που μας είπατε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα μιλήσατε για το 2050. Όμως οι γεωργοί έχουν να αντιμετωπίσουν τους αριθμούς που αναφέρει η οδηγία περί νητρικών αλάτων και πάρα πολλές χώρες όπως η Γερμανία καλούνται να εφαρμόσουν αυτήν την οδηγία. Ε, εσείς ε, μιλάτε για την ε, γεωργία συντήρησης που προφανώς και καλό θα ήταν να την εφαρμόσουν όλη η γεωργία, όμως οι πολιτικοί εκπέμπουν άλλα μηνύματα και ερωτώ Τελικά πώς θα τα καταφέρετε, ε, πώς θα καταφέρετε να πείσετε τους γεωργούς, μιλώ για την Ολλανδία και για άλλες χώρες. Οι γεωργοί ξέρετε προσαρμόζονται, αλλά πολλές φορές αυτά που λένε οι πολιτικοί είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή ήταν και η τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, την κυρία Ρεμότσα. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Η πολιτική έχει τεράστια ισχύ και μπορεί να το καταφέρει, αλλά η πολιτική χρειάζεται ένα χρόνο χάραξη και σχεδιασμού. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για μια μεγάλη επικράτεια όπω είναι αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τέτοια πολυμορφία, με διστάμενε απόψει πολλέ φορέ. Και εγώ προέρχομαι από μια οργάνωση που ασκεί πίεση. Ε, γι' αυτό και μίλησα για ένα τόσο μακρινό χρονικό ορίζοντα το 2050. Θέλω να είμαι ρεαλίστρια και να μην ζητάω εδώ ουτοπικά πράγματα. Δεν είμαι θεροβάμων. Δεν πρόκειται να ζήσουμε με όνειρα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως, να σημειώσουμε πρόοδο. Γι' αυτό ε, και ζήτησα και αυτό ήταν και το μήνυμα της ομιλίας μου. Τώρα σχεδιάζουμε τις μελλοντικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Λέω ότι με αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς νέες πολιτικές ώστε να έχουμε μια ολοκληρώση και να συμπεριλάβουμε και άλλες πτυχές. του νέους για παράδειγμα. Και βλέπουμε υπάρχει, ότι υπάρχει αλληλεμπίδραση τη γεωργία με άλλου τομεί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα περιλάβουμε στη γεωργική μα πολιτική να είναι όσο το δυνατό πιο ανοιχτή γίνεται απέναντι σε αυτή την πολυμορφία. Ήδη γίνονται κάποιε προσπάθειες, γι' αυτό και σα ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε προ αυτή την κατεύθυνση του ανοίγματο. Αυτά, ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Τορεμότσα και σα ευχόμαστε καλό ταξίδι μια και θα πρέπει να φύγετε. Καλό σα ταξίδι. Σας ευχαριστούμε και περνάμε στον τελευταίο μας εμπειρογνώμονα, τον κύριο Έκτορ Μολίνα Φάμπρα, καθηγητής γαστρονομίας. Έχετε και εσείς 10 λεπτά, κύριε Φάμπρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή Γεωργίας για την πρόσκληση. Νιώθω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και άκουσε τρεις κορυφαίες εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό. Εγώ είμαι καθηγητής βέβαια όπως με παρουσιάσατε, αλλά ταυτόχρονα είμαι και γεωργός και είναι το βιοποριστικό μου επάγγελμα η γεωργία. Από αυτό ζω. Δεν είμαι απλός καθηγητής. Και μάλιστα έχουμε ένα από τα σχέδια που δυστυχώς δεν μπόρεσα να σας το παρουσιάσω. Αυτό το παρουσίασα το 2012 νέο Γεωργό στο Φόρουμ Νέων Γεωργών, πρόκειται για ένα σχέδιο που στόχο έχει να αφήσει ένα περίγυρο υγιή ε, και καθαρό για εμά, του παραγωγούς και για την κοινωνία μας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θέλει να μειώσει στο έπακρο την ε, κατανάλωση νερού, κάνοντας καλύτερη αξιοποίηση του εδάφους ε, και συμβάλλοντας στην προσαρμογή των φυτών. Έτσι, ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε κάποιους επιβλαβείς ε, οργανισμούς των φυτών και να αξιοποιήσουμε και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εμείς έχουμε καταφέρει να ελέγχουμε κάθε καλλιέργεια σχεδόν και από το σπίτι μας μερικές φορές. Πρόκειται για ένα πολύ υπεύθυνο project και μάλιστα με μεγάλη ηθική και διοντολογία. Γιατί αυτό μας προβληματίζει πάντα. Τι κάνουμε στο σχέδιό μας. Ή ε, μάλιστα το σχέδιό μας δεν έχει λάβει καμία επιδότηση, καμία ενίσχυση, στηρίζεται 100% στο ιδιωτικό ε, κεφάλαιο και προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό που ακριβώς συζητάτε εσείς σήμερα, τα συστήματα καλλιέργειας, να βελτιώσουμε την παραγωγή, προς όφελος όμως του πλανήτη μας και προς όφελος του περιβάλλοντός μας. Γιατί Βέβαια, δυστυχώ ακόμη δεν λαμβάνουμε καμία επιδότηση, καμία ενίσχυση δημόσια. Στηριζόμαστε 100% στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Και μια και μιλούμε για γεωργία, χαίρομαι που είμαι ο τελευταίο ομιλητή, γιατί πρόλαβα να ακούσω του προηγούμενου και να προσαρμόσω ανάλογα και τη δική μου ομιλία. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και αυτά που είδαμε. Ακούσαμε τα σχόλια για την γλυφωσάτη που χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις. Ε, μιλήσαμε και για άλλα προϊόντα και είπαμε πολλά και ακούσαμε πολλά για τη Γεωργία. Έχουμε το 2016 όμως κάτι που ακόμη δεν αναφέρεται. Μία λέξη που θα πρέπει να την αναφέρουμε πολύ πιο συχνά, τη λέξη υγεία. Γιατί ζούμε σε μία πολύ πλούσια ήπειρο, ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί το 1 τέταρτο του πληθυσμού θα υποφέρει από καρκίνο. Και όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας ε, αντιμετωπίζουν καρκίνο, αντιμετωπίζουν διαβήτη, το διαβήτη τύπου 2, που μάλιστα παρόλο που ήταν καταρχήν ο διαβήτη των ενηλίκων, αρχίζουν και τον αντιμετωπίζουν και παιδιά. Αντιμετωπίζουμε καρδιακέ παθήσει, πολλά σοβαρά προβλήματα υγεία, παρόλο που ζούμε σε εύπορε χώρε, σε πλούσιε χώρε, σε, ένα πλούσιο, σε μια πλούσια ήπειρο. Μάλιστα, πριν έρθω, προβληματιζόμουν με διάφορα ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι θα πει Ευρώπη και μάλιστα έψαξα στο, στην πύλη 3 3W www.europa.eu που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικονομική και πολιτική ένωση ε, ιδιόρυθμη που στηρίζεται στην ε, πρόθεση της οικονομικής συνεργασίας που στο μέτρο που αυξάνεται η οικονομική ελεξάρτηση μεταξύ των χωρών μειώνονται οι πιθανότητες σύγκρουσης. Πρόκειται για μια ενιαία μεγάλη αγορά που ε, στόχο έχει να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό του. Αυτά λέει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πύλη Ευρώπα ΕΟΥ. Που, τι σημαίνουν όλα αυτά, δηλαδή να καταφέρουμε οι Βέλγοι να σκέφτονται ως Ισπανοί, οι Ισπανοί να σκέφτονται σαν τους Ολλανδούς, οι Ολλανδοί σαν τους Πορτογάλους και υπάρχουν 700 και ε, συνδυασμοί, 700 και συνδυασμοί ώστε να καταφέρουμε ο ένας να σκέφτεται όπως ο άλλος και να υλοποιήσουμε το στόχο μας που είναι μια ισχυρή ένωση. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή που στηρίζεται στην καλλιέργεια σπεριδοειδών. Εκεί όμως ε, τα άρθρα του τύπου λένε ότι οι Βρυξέλλες ε, ανοίγουν τις πόρτες ε, στα πορτοκάλια της Νοτιού Αφρικής ή μειώνουν τους δασμούς ε, για τα πορτοκάλια της Νότιας Αφρικής ή θέτουν σε κίνδυνο τις ε, ισπανικές και τις ιταλικές ποικιλίε σπεριδοειδών ή οι Βρυξέλλες επιτρέπουν στο Μαρόκο να εξάγει 475.000 ε, τόνους εσπεριδοειδών και μάλιστα αδασμολόγητων. Αυτά είναι που βλέπουμε στον τύπο τον τοπικό. Αυτό δεν έχει σχέση με τη σημερινή δημόσια κρόαση. Αλλά όταν ε, μία περιοχή όπως η δική μου όπου είδε να έρχονται πριν από πάρα πολλά χρόνια τα πρώτα μανταρίνια από την Κίνα και που εξακολουθεί να είναι παγκόσμια δύναμη στην παραγωγή και εξαγωγή περιδοειδών, ακούγοντας τέτοιες ειδήσει. Ε, μας ε, οδηγούν σε πολύ δυσάρεστα και απογοητευτικά αποτελέσματα. Έχουμε ήδη 25% ε, μείωση των καλλιεργιών των εσπεριδοειδών και 20% απερίμωση της, ε, των ισπανικών εδαφών. Κάτι τέτοιο φυσικά απογοητεύει και αποθαρρύνει την ισπανική κοινωνία. Επίσης, θα ήθελα να σκεφτούμε τι, τι σημαίνει γεωργός. Εγώ σας είπα ότι εγώ προσωπικά είμαι γεωργός και οι ε, γονείς μου και οι παππούδες μου ήταν γεωργοί. Τι έκαναν οι γεωργοί. Οι γεωργοί δημιουργούσαν ένα ευτυχισμένο περίγυρο. Ε, ήταν παραγωγή και μάλιστα στην γενέτειρά μου είχαμε επώνυμες ντομάτες, δεν είχαμε ντομάτες άνοστες ή είχαμε επώνυμα ροδάκινα, όχι ροδάκινα χωρίς γεύση. Ή όσοι είστε οπαδοί, λάτρεις της παέγια, θα ξέρετε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο φασόλι, φασόλι λίμας που χρησιμοποιούμε. Το 90% των φασολιών λίμας το εισάγουμε στην Ισπανία από την Αμερική. Και έτσι δίνουμε έμφαση στις ξένες παραγωγές από ό,τι στην κατανάλωση ντόπιων προϊόντων. Το έργο του Γεωργού είναι ένα έργο αξιοπρεπές που διαφυλάσσει και διατηρεί το περιβάλλον και στο Γεωργό εμπιστευόμαστε την υγεία μας. Παρόλο που όπως σας είπα προηγουμένως όλο και, απειλεί, όλο και απειλείται στη σύγχρονη εποχή. Εγώ είμαι κάτω των 40 ετών, άρα με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε νέος Γεωργός. Το 1979 πάνω από το 20% των γεωργών ε, ήταν νέοι κάτω των 35 ετών. Σήμερα είναι 5,7% μόνο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από 30% είναι πάνω των 65 ετών. Δεν έχουμε δηλαδή πολλούς νέους γεωργούς. Γιατί σήμερα μιλήσαμε για διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους. Αλλά τι γεωργία περιμένουμε αν έχουμε ένα γυράσκοντα αγροτικό πληθυσμό. Αν δεν κάνουμε μια πραγματικά καμπή, μία στροφή 180 μοιρών, ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικές θέσεις απασχόλησης, γιατί ταυτόχρονα διανύουμε μία σοβαρή κρίση και έχουμε προβλήματα και θέσεων απασχόλησης και κυρίως αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης. Αν δεν κάνουμε λοιπόν μία σημαντική στροφή, τότε θα έχουμε μία γεωργία με ημερομηνία λήξης, δυστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπε και η σας, ε, εμείς προσπαθούμε να ανακτήσουμε και παλιές ξεχασμένες ποικιλίε, παραδοσιακές, προσαρμόστες σε συγκεκριμένο περιβάλλον και επίσης ε, ε, καλλιέργειες που χρειάζονται λιγότερο νερό. Αυτή τη στιγμή 60% των ε, παγκόσμιων σπόρων τις ε, μονοπολούν 6 με 8 επιχειρήσεις. Ενώ πριν από μερικά χρόνια ήταν χιλιάδες οι επιχειρήσεις που είχαν τον παγκόσμιο έλεγχο των ε, σπόρων. Το ίδιο ισχύει και με τα φυτοφάρμακα και τα ζυζανιοκτώνα. Σχεδόν υπάρχει ε, απόλυτο μονοπόλιο και απόλυτο μονοπόλιο των γενετικών τροποποιημένων οργανισμών που ε, τους λιμένονται οι πολυεθνικές. Και οι υπόλοιποι γεωργοί είναι υποδουλωμένοι, είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν από συγκεκριμένη πολυεθνική που έχει το δίπλωμα βρεσιτεχνίας ε, τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Στη Βαλένσια το 2013 ανακαλύψαμε ένα φυτοφάρμακο, το τερμπουμετόνα ντεσετήλ και μάλιστα 10 χρόνια μετά την απαγόρευση της χρησιμοποίησής του εμφανίστηκε στο νερό της Βαλένθια ε, και σε μια πόλη 45.000 κατοίκων. Και μάλιστα ο ποταμός Χούκαρ που άρδευε εκατοντάδες χιλιάδες καλλιέργειες ε, ήταν μολυσμένο από αυτό το φυτοφάρμακο. Και επαναλαμβάνω, 10 χρόνια μετά την απαγόρευσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν ακόμη σημαντικά υπολείμματα αυτού του φυτοφαρμάκου στη Βαλένσια. Και μάλιστα ε, έχουμε κατασπατάληση τροφίμων. 700 κιλά το χρόνο ε, ανακάτοικο ε, πετάμε τρόφιμα. Και επισης 35% ε, των τροφίμων ε, τα μετατρέπουμε σε απόβλητα. Και έχουμε και μεγάλη κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακα. Βλέπετε τι αντίκτυπα έχουν όλα αυτά για τον παραγωγικό μας ιστό. Επιπλέον, εφαρμόζουμε ένα βιομηχανικό μοντέλο που έχει φτάσει πια στα όρια του εξαιτίας της θέρμανσης του πλανήτη που βρίσκεται στους πηχαίους τίτλους όλων των ε, εφημερίδων εξαιτία ε, της μονοκαλλιέργειας και της διάβρωσης του εδάφους, εξαιτία της ατμοσφαιρικής ρύθμις, ε, ρήπανσης, εξαιτία της των υδάτων, της θάλασσας, των ωκεανών και των γλυκών υδάτων. Έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και επίσης είμαστε υποδηλωμένοι στον έλεγχο των πολυεθνικών. Όλα αυτά είναι τα προβλήματά μας. Τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε. Ως πολίτης, το μόνο που θα μπορούσα ε, να σας παρακαλέσω, γιατί σας δίνουμε την ψήφα μας και άρα την εμπιστοσύνη μας, είναι από εσάς μια δέσμευση, μια δεντολογία, μια ηθική, μια επιθυμία να αλλάξουμε αυτή την στραβή κατεύθυνση που πήραμε. Γιατί οι αλλαγές, όπως είπε η κυρία από την Ολλανδία, θα πρέπει να γίνουν αργά, αλλά το θέμα είναι να μην χάνουμε χρόνο. Και όπως είπε και ο Λεωνάρδο Μπός, μια κοινωνία Λεωνάρντο μια κοινωνία που αποφασίζει να οργανωθεί χωρίς ελάχιστη ηθική, χωρίς αλτουρισμό και χωρίς σεβασμό στη φύση, χαράζει το δρόμο προς την αυτοκαταστροφή της. Αυτά είπε ο Λεωνάρντο Μποφ, που θαυμάζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, λίγος χρόνος μας έχει μείνει, οπότε παρακαλώ πολύ σύντομε ερωτήσεις. Κύριε Άγνιου, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι ο μιλητής ζήτησε λύση. Θα του δώσω μια λύση αν ε, προσπαθήσετε να κάνετε κάτι, έχουμε επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν χρησιμοποιήσει ε, μεθόδους καλλιέργειας φυτών που μπορούν να δώσουν. Βεβαίως έχουμε νέες ε, τεχνικές που έχουν καταδικαστεί από αυτό το κοινοβούλιο. Θα σας δώσουν όμως μια μείωση χρήσης ενέργειας, μείωση στην διάβρωση, μείωση στην χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων αλλά όλοι λένε δεν πρόκειται να πλησιάσουμε αυτές τις μεθόδους μέχρι ότου υποστηρίξουμε ε, τους επιστήμονες μας ε, στις ε, καινοτομίες. Αν εξακολουθήσουμε να τους λέμε ότι είναι ανοησίες, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ. Δεν θέλει άλλο κανείς το λόγο, οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Φάμπρα για την απάντηση. συγγνώμη, κύριο Ντε, μια σύντομη ερώτηση επίση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και για την εισήγησή σας. Αλλά τώρα, το τι σχέση έχει αυτή η εισήγηση με μεθόδους ε, συντήρησης ε, γεωργίας, ε, εγώ δεν το κατάλαβα. Ίσως θα πρέπει αυτά που μας είπατε να τα πείτε σε άλλες, σε άλλα φόρουμ, γεωλογικής, φύσης, οτιδήποτε άλλο και εδώ να μας πείτε για θέματα που μας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ σύντομα οι απαντήσει. Sí, volviendo eh, Ως προς τη δεύτερη παρέμβαση. Εγώ σας μίλησα για τα αίτια του κακού, τα αίτια του προβλήματος που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Όπως σας είπα, εγώ δεν ήρθα εδώ για να σας δώσω λύσεις. Μπορώ να συμβάλλω στην αναζήτηση λύσεων. Αλλά αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι σε τι περιβάλλον ζούμε σε τι περίγυρο ζούμε, πού πού κινείται η κοινωνία μας και τι μόλυνση έχουμε σε όλα σχεδόν τα επίπεδα εδαφών, ατμόσφαιρας, νερού. Σας είπα ότι εμείς εφαρμόζουμε μία γεωργία που σέβεται το περιβάλλον, σέβεται το περίγυρο. Δεν κάνουμε άρρωση και μπορώ να σας μιλήσω για την μεθοδολογία και το σύστημα που εφαρμόζουμε στην, στις καλλιέργειές μας. Χρησιμοποιούμε τη μηδενική άρρωση. Επίσης, ε, ε, προσφέρουμε τρόφιμα στα παιδιά με πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και διαχειρίζονται σωστά το έδαφος. Το μήνυμά μου μπορεί να μην ε, πρότεινε λύσεις. Και όπως είπατε, ίσως θα ήταν κατάλληλη με τέτοια παρέμβαση σε άλλου είδου ομίγυρη. Αλλά όπω σα είπα, εγώ δεν ήθελα να φέρω λύσει, αλλά να συμβάλλω σε μια συνειδητοποίηση, σε μια αφύπνιση τη συνείδησης τη κοινωνία. Καλώ, εντάξει, δεν είχαμε... Ήταν μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο γεωργών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολύ σύντομη παρέμβαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. E Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο για να σα υπενθυμίσω ποια είναι βασικά τα εργαλεία τη κοινή γεωργική πολιτική, ποια εργαλεία έχουμε στα χέρια μα και πώ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποιε απόψει ε, που παρουσιάστηκαν σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να επενθυμίσω ότι η πολιτική γεωργική ανάπτυξη περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα μέτρα ε, προστασία του περιβάλλοντος που θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε κάποιες από τις τεχνολογικές ε, λύσεις ε, κάποια από αυτά που αναφέρθηκαν. Θα ήθελα όμως να επενθυμίσω ότι ε, όσον αφορά το δίκτυο για την ε, γεωργική ανάπτυξη τα μέτρα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και θα πρέπει να εργαστούμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα επίση να σα υπενθυμίσω ότι το σύστημα το European Innovation Partnership, αυτό το σύστημα εταιρικών σχέσεων και συνεργασιών για τη Γεωργία, αυτό έχει καταλήξει σε κάποια έγγραφα τα οποία έγγραφα αυτά είχαν ιδιαίτερα θετική, πολύ καλή επίχυση από πλευράς γεωργών. Και θέλω επίσης να επενθυμίσω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες ομάδες που δημιουργούνται, οι οποίες ομάδες πραγματικά μπορούν να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στη διάδοση αυτής της τεχνολογίας. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω και κάποιες ερωτήσεις ε, πριν ε, κλείσω. Δηλαδή θέλω να ε, ρωτήσω γιατί δεν βρίσκω απαντήσεις. Το 10% των εκπομπών προέρχονται από το έδαφος. Ε, είναι Τώρα, οι γεωργικές εκπομπές ποιο ποσοστό καταλαμβάνουν σε αυτό το 10%. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εμβαθύνουμε στο τι σημαίνουν όλες αυτές οι τεχνικές κάτω από το πρίσμα ε, της απόδοσης για τον Γιώργο. Μιλήσαμε για μείωση των δαπανών κατά 19%. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά για τον Γιώργο ε, όσον αφορά κυρίως το εισόδημά του. Αυτές είναι νομίζω σημαντικές ερωτήσεις. Και τέλος ε, θέλω να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε όπως το έκαναν ίσως και οι συγητές, να κατανοήσουμε τι κοστίζει σε επίπεδο οικονομίας. Αυτό είναι ερώτηση κλειδί. Ε, τόνο τόνος ε, άνυδρου άνθρακα που κατορθώνει κανείς να δεσμεύσει στο έδαφος, ποιο είναι το κόστος αυτής της δέσμευσης άνθρακα. Γιατί νομίζω και αυτό είναι καθοριστική σημασία από πλευράς πολιτικής. Έχω πρόβλημα γιατί για πρώτη φορά ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέτει ερωτήσει. Συνήθω απαντούσε απαντούσες ερωτήσει. Και τώρα για πρώτη φορά, αυτό είναι άνευ προηγουμένου, βλέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέτει ερωτήσει. Σα ευχαριστώ. Έχουμε μια νέα ποιότητα εδώ σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν κάποιο είναι σε θέση να δώσει έστω και σύντομη απάντηση, θα ήμουν ευγνώμων. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω, κυρία εμπειρογνώμων, γιατί πρέπει να πάμε και στην άλλη συνεδρίαση. Ναι, πάντως θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο για τη δέσμευση άνθρακα σε σχέση με την γεωργία συντήρησης, να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί και προσεκτική όταν μιλάμε, ε, όταν λέμε ότι μειώνεται η αλλαγή ε, του, του κλίματος ε, με την δέσμευση και αποθήκευση στο έδαφος του άνθρακα. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το πει, αλλά υπάρχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο πάνω στρώμα, αλλά στο βάθος του εδάφου σαν εκτάριο δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο απόθεμα ε, άνθρακα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα και οι επιστήμονες συμφωνούν ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί σχετικά με τα πλεονεκτήματα της δέμευσης άνθρακα στην γεωργία συντήρησης. Βεβαίως μειώνονται οι ε, οι εκπομπές από τα καύσιμα και βεβαίως έχουμε τα νητρικά άλατα και έχουμε επίσης και άλλα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν υπάρχει λοιπόν απλή απάντηση, δεν μπορώ να σας μιλήσω για την αξία της δέσμευσης άνθρακα στην γεωργία συντήρησης. θα είμαι λακωνική. Θα ήθελα απλώ να σας υπενθυμίσω κάποια στοιχεία που έχουμε από μελέτες σχεδίων. Και στα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι η δέσμευση άνθρακα στο, του εδάφους ήταν 20 πλάσια σε σχέση με τη μείωση που γίνεται από την μηδενική άρρωση. Αυτό έδειξε το σχέδιο Life Plus agri Park που έγινε στην Ισπανία. Βέβαια και η επιστήμη μα λέει ότι πολλέ φορέ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να τα βλέπουμε όλα αυτά με προσοχή. Αυτά ολοκληρώνεται αυτό το τμήμα τη συνεδρίαση. Θα πρέπει να αλλάξουμε αίθουσα τώρα. Ήταν ενδιαφέρουσα πολύ δημόσια αυτή ακρόση εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας και θα τις αξιοποιήσουμε και στο μέλλον αυτές τις πληροφορίες που λάβαμε. Επαναλαμβάνω, η συνέχεια στην αίθουσα 1G3 στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. 1G3 αμέσως τώρα. Και ευχαριστώ και πάλι θερμά τους καλεσμένους μας.